ladies and gentlemen, dear colleagues, a warm welcome. Συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Ένα θερμό καλωσόρισμα. Είναι 4 και 8. Να ξεκινήσουμε τη σύντομη συνεδρίασή μας για σήμερα. Ε, ως προς την ημερήσια διάταξη, να διευκρινίσω ότι το 7, η ανταλλαγή απόψεων με τον Ζωάο Αλμέιντα, που είναι ο επιτετραμένο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέσβη του το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αναβληθεί, γιατί έχει ανελημμένε υποχρεώσει στο Λονδίνο. Σε μεταγενέστερη ημερομηνία λοιπόν θα γίνει αυτή η συνάντηση και σε ό,τι αφορά τι πρόσφατε εξελίξει στην Λιβύη και την σύνοδο χθε στο Βερολίνο θα προσθέσουμε το 11β για το θέμα αυτό. Ανταλλαγή απόψε με τον κύριο Τζεντιλίνη, εκτελεστικό διευθυντή για τις σχέσεις με την Μέση Ανατολή, την Μορεφρική και υπεύθυνο τη ε, Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Αύριο το πρωί θα τον δούμε και θα πάει η συνεδρίαση μας μέχρι τη μία. Συμφωνείτε? Ωραία. Εγκρίνεται λοιπόν η μερίσια διάταξη. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Μία ανακοινώση έχω να κάνω. Εάν κάθεται κανείς εδώ στο Προεδρείο και όταν έχουμε προσκεκλημένους, είναι πολύ ενοχλητικό αυτή η πόρτα να βροντάει κάθε 30 δευτερόλεπτα. Δεν μπορεί κανείς να συγκεντρωθεί και ενοχλεί και τους ομιλητές να μπαινοβγαίνουν συνέχεια διάφοροι. Θα ζητήσω λοιπόν αυτή η πόρτα να κλείσει και να μπαίνουν όλοι από την άλλη είσοδο για να γίνεται λιγότερο θόρυβος. Δεν είναι ευχάριστο για τους προσκεκλημένου μας. Ρακέλ, για τους προσκεκλημένου μας έχουμε αυτή τη στιγμή κάποιον. Ωραία λοιπόν, θα μπαίνετε από το πλάι, νέος κανόνας. Ε, Θα προσκαλέσετε τους αντιπροέδρους. Ε, κοιτάξτε, μπορεί να μπορούσα να σας πω περισσότερα για τους αντιπροέδρους. Το έχω συμπεριλάβει στην αμυρίσια ε, ε, διάταξη των συντονιστών που θα ξεκινήσει στις 6.30. Αλλά παρακαλώ να ενημερώσετε τις τρεις ομάδες που έχουν ε, σχέση με το θέμα αυτό, διότι πρέπει να βρούμε μια λύση Γι' αυτό ακριβώ έχουμε τους αντιπροέδρους στις επιτροπές. Μπορούμε να βρούμε κάποια κυρία από αυτέ που είναι υπεύθυνε στις τρει ομάδε. Κάτι πρέπει να γίνει. Αλλά θα το συζητήσουμε στο επίπεδο των συντονιστών, κύριε Μπασέσκου, στο... στους συντονιστές που αρχίζουν σε μισή ώρα. Στο μεταξύ, Εάν αυτή η Επιτροπή δεν μπορέσει να εκλέξει αντιπροέδρους, θα ζητάμε να προεδρεύουν με σειρά αρχαιότητας. Οι συνάδελφοι, αυτή είναι η μόνη λύση. Διότι... Ρέινολ, το ξέρω ότι και σε έχει υπηρετήσει πολύ καιρό, αλλά υπάρχουν και άλλοι. Οι 7 παλιότεροι είναι από το ΕΛΚ. Ούτε αυτό γίνεται και είναι και όλοι άντρε. Δεν είναι λύση. Θα τα ξανασυζητήσουμε και μετά. Τρία λοιπόν. Ανακοίνωση Προέδρου βάσει του άρθρου 214 του ιστορικού κανονισμού το, ε, τα, αρχή, πρακτικά των αποφάσεων των συντονιστών 4 Δεκεμβρίου, 9 και 10 Ιανουαρίου βρίσκονται στον ιστότοπο της ΑΦΕΤ και τον έχετε, έχετε στο φάκελό σας με τα υπόλοιπα εγγραφά της σημερινής συνεδρίασης. 4. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων 6 και 7 Νοεμβρίου και 25 Νοεμβρίου. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Ας εγκρίνουμε χωρίς αλλαγές τα πρακτικά. Και μετά πάμε στο 5 Πρώτη εξέταση του σχεδίου γνωμοδότηση για τη σύναψη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Δημοκρατία τη Λευκορωσία για την επανεισδοχή ε, πολιτών που κατοικούν ε, χωρί εξουσιοδότηση. Κύριε Στραβίτσιου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι είναι μια συμφωνία αυτή μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας όσο είναι ακόμα δημοκρατία. Ελπίζω να παραμείνει το όνομα αυτό και ο τίτλος αυτός και η ίδια ιδιότητα ε, στο μέλλον. Αυτές οι δύο συμφωνίες και θα ήθελα να παρουσιάσω και τα δύο σχέδια γνωμοδότησης και τις δύο εκθέσεις, γιατί έχουν να κάνουν με παρεμφερή αντικείμενο, αντικείμενα το ένα πλαισιώνει το άλλο. Αυτές οι δύο συμφωνίες λοιπόν εμπίπτουν ακολουθούν την πρωτοβουλία της εταιρική ε, σχέσης προς τα ανατολικά, την ανατολική εταιρική σχέση, η οποία, ε, την οποία γιορτάσαμε πέρσι ε, διότι έκλεισαν τα 10 χρόνια από την ανάληψη της πρωτοβουλίας αυτής. Έχουμε λοιπόν ε, τη Συμφωνία Επανεισδοχής και τη διευκόλυνση για την έκδοση θεωρήσεων. Ε, πρέπει να σας πω, συναδελφοί, ότι η Λευκορωσία είναι η χελώνα, αν θέλετε, στην ανατολική εταιρική σχέση. Είναι η χώρα που προχωρά με τον πιο βραδύ ρυθμό, δεν έχουμε μέγιστα επιτεύγματα ως προς τα θέματα που μας απασχολούν. Ωστόσο, από τη Συμφωνία του Συμβουλίου από το Φεβρουάριο του 2011. Τελικά χρειάστηκε τρία χρόνια για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις το 2014 και πέντε χρόνια μας χρειάστηκε για να καταλήξουμε σε αυτές τις δύο συμφωνίες για την επανεισδοχή και την ε, διευκόλυνση για την έκδοση θεωρήσεων. Και μία κάποια πρόοδος έχει σημειωθεί σε ό,τι έχει να κάνει με τα νομικήστικά τα νομικά και τυπικά ε, ζητήματα των συμφωνιών αυτών. Δεν έχει κλείσει οριστικά καμία από τις δύο συμφωνίες με τη δημοκρατία της Λευκορωσίας. Και δεν χρειάζεται να σας πω ότι ένα πλουστευμένο καθεστώς κινητικότητας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της δημοκρατίας της Λευκορωσίας τελικά τι θα κάνει, θα ενισχύσει την επαφή την επικοινωνία μεταξύ των πολιτών, μεταξύ των ανθρώπων και αυτό είναι δικό μας προσδοκόμενο, είναι κάτι που στηρίζουμε, είναι κάτι που μπορεί να παράγει περισσότερα αποτελέσματα και να οδηγήσει σε μεγαλύτερη διάδραση, σε μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ ημών και πολιτών της Λευκορωσίας. Οφείλω να αναγνωρίσω ότι η πολιτική κατάσταση στη χώρα αυτή παραμένει ιδιαίτερα περίπλοκη. Και στις πρόσφατες εκλογές του Νοεμβρίου του 2019 ε, ε, ε, έδωσαν λαβή για πολύ σημαντικές παρατηρήσεις και κριτικές από τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και άλλους οργανισμούς και πρέπει να πω ότι τα διεθνή πρότυπα για τις οικουμενικές θεμελιώδεις ελευθερίες και για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, δεν τηρούνται στο 100% παραμένουν κενά εκεί και σφάλματα. Η αξιωματική αντιπολίτευση συνεχίζει να υφίσταται πιέσεις από το καθεστώς που έχει τα ενία της εξουσίας στο Μίνσκ. Ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλω να πω, συνεχίζουν να ε, επιδεικνύουν ένα κριτικό πνεύμα, ε, να ασκούν κριτική για την πολιτική της Λευκορωσίας όσον αφορά στο θέμα της πυρηνικής ασφάλειας και το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας το οποίο θα ολοκληρωθεί στη χώρα αυτή του επόμενους μήνες είναι η αλήθεια ότι δεν πληρεί τα υψηλότερα δυνατά ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. Όμως, με τη συμφωνία αυτή ενθαρρύνεται η επικοινωνία, η επαφή μεταξύ των πολιτών, μεταξύ των χωρών και για αυτούς τους λόγους πιστεύω ότι πρέπει να τη στηρίξουμε. Όχι μόνο τη συμφωνία για την επανεισδοχή, αλλά και τη συμφωνία για τη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων, της έκδοσης βίζας δηλαδή. Αυτά τα δύο συνοδεύει το ένα το άλλο, πορεύονται ταυτόχρονα για να δημιουργήσουν το απαραίτητο, το απαραίτητο πλέγμα νομικών προϋποθέσεων που χρειάζονται για να καλλιεργήσουμε περαιτέρω τη σχέση μας με τη χώρα αυτή. Ζητώ τη στήριξή σας, διότι η καθήκον της Επιτροπής μας είναι να συντάξει ένα σχέδιο γνωμοδότησης. Οι συνάδελφοί μας από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών είναι αυτοί που θα λάβουν και την τελική απόφαση. Και με αυτά θα ήθελα να ολοκληρώσω κάπου εδώ, κάπου εδώ απευθύνοντας αυτή την έκκληση προς τα εσάς να εγείρετε το ζήτημα του απολύτου σεβασμού, της απολύτου τήρησης των θεμελιωδών ελευθεριών, των οικουμενικών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ε, να ε, στη Λευκορωσία, να μην μπορούν μόνο οι πολίτες αυτοί να ταξιδεύουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να μπορούν να αξιοποιήσουν και να απολαύσουν όλες αυτές οι ελευθερίες και όλα αυτά τα δικαιώματα που έχουμε εμείς στην Ευρώπη και εντός των συνόρων της δικής τους χώρας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτών των σημείων του 5 και του 6, οπότε θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους να τοποθετηθούν και για τα δύο θέματα. Πάμε στους Κιώδης. Η Σάντα Κανιέτε έχει πρώτη το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Αστρεβίτσιους, για τις δύο αυτές γνωμοδοτήσεις απαιτήσει τις οποίες στηρίζω με όλη μου την καρδιά. Η χορήγηση καθεστώτος διευκόλυνσης έκδοσης θεωρήσεων αποτελεί το πρώτο βήμα προς την πλήρη απελευθέρωση των θεωρήσεων που απολαμβάνουν αυτή τη στιγμή οι πολίτες της Γεωργίας, Μολδαβίας και της Ουκρανίας. Επίσης είμαι υπέρ της ενίσχυσης των διαπροσωπικών επαφών που αναφέρατε. Είναι σημαντικό αυτό λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης όπου η αντιπολίτευση στη Λευκορωσία ε, υφίσταται καταστολή και καταπίεση ενώ δεν υπάρχουν, ε, δεν διεξάγονται ελεύθερες ε, δημοκρατικές εκλογές. Παρά τις ε, συστάσεις του ΑΣΕ και άλλων οργανισμών και παρά τις συναντήσεις και συνεδριάσεις που είχαμε και εμείς ως ευρωβουλευτές με τις λευκορωσικές αρχές. Θετικό είναι το γεγονός ότι πρόκειται για ένα στρατηγικό βήμα για να μειωθεί και η ρωσική επιρροή στη Λευκορωσία. Οι προσπάθειε της Μόσχας για την αναβίωση μιας ένωσης μεταξύ Ρωσίας και Λευκορωσίας έχει κάνει ορισμένους παρατηρητές να πούν ότι αυτό, ένα τέτοιο βήμα, μια τέτοια προοπτική θα ε, μείωνε ε, μεγάλο μέρος της ανεξαρτησίας της Λευκορωσίας. Υποστηρίζω λοιπόν εγώ αυτές τις δύο γνωμοδοτήσεις και το ίδιο καλό και τους συναδέλφους να κάνουν. Ευχαριστούμε Σάνδρα Κανιέτε, σοσιαλιστές. Ο Σιώδης είναι ο κύριος Νόιζε, αλλά δεν είναι εδώ. Ίσως θα ήθελε κάποιος άλλος το λόγο εκ μέρους των σοσιαλιστών. εκ μέρους των Πρασίνων η κυρία Τόμπαντελ. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς οι Πράσινοι υποστηρίζουμε το μηχανισμό, την Συμφωνία Διευκόλυνσης Χορήγησης Θεωρήσεων. Όμως δεν συμφωνούμε με την διασύνδεση αυτού του θέματος με την ε, συμφωνία για την επανεισδοχή. Γενικά πάντως η άποψή μας είναι ότι πρέπει να διευκολυνθεί η χορήγηση θεωρήσεων γιατί όπως είπε και η Σάντρα είναι πολύ σημαντικές οι διαπροσωπικές επαφές μεταξύ των ανθρώπων Ιδίω ε, μεταξύ φοιτητών, απλών πολιτών, ανθρώπων, πρέπει να έχουν οι άνθρωποι αυτοί την ευκαιρία να εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να λαμβάνουν θεώρηση Σέγγεν με πιο εύκολο, απλοποιημένο τρόπο από ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Γνωρίζουμε ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν εμπειρία από πρώτο χέρι για το τι θα πει ζωή εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Σάνδρα ανέφερε επίσης και τις προσπάθειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας να επιχειρήσει, εν πάση περιπτώσει, να κινηθεί προς μια επανένωση ε, με την Λευκορωσία στο πλαίσιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Οπότε είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λευκορωσίας έχει βελτιωθεί, οι σχέσεις έχουν βελτιωθεί και από αυτή την άποψη υποστηρίζουμε και εμείς τη γνωμοδότηση αυτή. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κυρία Μαριανή, θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ομάδα μας βεβαίως θα στηρίξει αυτές τις δύο συμφωνίες. Είμαστε θετικός διακείμενη. Έχω παρακολουθήσει το θέμα της επανεισδοχής σε Εθνικό Κοινοβούλιο, στο Γαλλικό Εθνικό Κοινοβούλιο. Η Λευκορωσία ήταν μια χώρα η οποία συνεργαζόταν άψογα και δεν είχαμε ποτέ προβλήματα επανεισδοχής. Τώρα για τη Συμφωνία για τη Διευκόλυνση Θεωρήσεων. Συμφωνούμε όλοι όντω, η καλλιέργεια της δημοκρατίας καθίσταται δυνατή διευκολύνοντας τις ανταλλαγές παντός είδους. Άρα στηρίζουμε αυτή τη Συμφωνία Απλούστευσης για τις θεωρήσεις. Οφείλουμε όμως να διατυπώσουμε την εξή παρατήρηση. Χρειάστηκαν πάρα πολλά χρόνια για να υπογραφεί η συμφωνία και ορθά και καλώ το έθεσε αυτό και το είπε αυτό ο εισηγητή. Δεν ξέρω ποιο έχει την ευθύνη, η ευρωπαϊκή πλευρά ή η πλευρά τη Λευκορωσία. Εδώ και πολλού μήνε θα μπορούσαμε να είχαμε υπογράψει τη συμφωνία, πολύ νωρίτερα δηλαδή. Άρα τίθεται το ερώτημα τη τιμή ε, για την έκδοση των θεωρήσεων. Και αν δεν απατώμε, η τιμή, το κόστο δηλαδή, αυξάνεται από τι 2 Φεβρουαρίου. Ο πρέσβη τη Λευκορωσία είχε ζητήσει, ε, είχε παρεύει πριν από την ε, υπογραφή και είχε ζητήσει να παραμείνουμε στα 60 ευρώ που είναι, ήταν η τιμή ε, όταν είχε ξεκινήσει η συζήτηση, κοιτάξτε, 20 ευρώ για μας δεν είναι τίποτα, αλλά 20 ευρώ για έναν φοιτητή από τη Λευκορουσία είναι ένα τεράστιο ποσό. Από τα 60 να ε, πάει 20 ευρώ παραπάνω. Επομένως, στηρίζω ε, στηρίζουμε τη συμφωνία και θέλουμε το κόστος να παγώσει στα 60 ευρώ και να μην αυξηθεί κατά 20 ευρώ. Αυτό ζητούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό όταν θα δώσουμε το λόγο στους ε, εκπροσώπους της Κομισιόν και στον συνάδελφο Πέτρας. Όμως ε, θα ήθελε πρώτα να πάρει κάποιο το λόγο από τους συναδέλφους του ECR. Όχι. Από την ΚΟΕ. E, επίσης όχι. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι. Έχουμε περισσότερους ομιλητές. Ο κύριο Γκάλα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Φυσικά υποστηρίζω και εγώ τις δύο αυτές προτάσεις. Και νομίζω ότι συμφωνούμε και πολιτικά. Αν το θέμα ήταν μόνο το καθεστώς ε, και να ανταμυφθεί αυτό, αυτό βεβαίως δεν θα έπρεπε να γίνει. Το είπε και η Πέτρα, πραγματικά οι εκλογές που ε, είδαμε να διεξάγονται τον Νοέμβριο στη χώρα ήταν οι από την δεκαετία του 90 και ε, διαπιστώσαμε και άλλες ε, περίεργε συμπεριφορέ, όπως και στις τελευταίες διαδηλώσει, ε, στις οποίες κατέβηκε η αντιπολίτευση εναντίον αυτών των προσπαθειών εκ μέρους Ρωσίας για προσέλκυση τη Λευκορωσία στο άρμα τη. Όμω είδαμε και άλλα φαινόμενα τα τελευταία χρόνια. Ο κύριος Πρένιτς από τους χριστιανοδημοκράτες ε, του επευλήθη ποινή 30 ημερών ε, κράτησης με αναστολή για συμμετοχή σε αυτές τις διαδηλώσεις. Ε, παρά το γεγονός ότι δεν έπραξε τίποτα το παράνομο. Οι διαδηλώσεις αυτές αφορούσαν την αναστολή, την την αναχέτηση μάλλον ε, των ε, ρωσικών ε, προσπαθειών για προσετερισμό της Λευκορωσίας. Οπότε και από άποψη υποστήριξης της αντιπολίτευσης είναι σημαντικό. Να πω κάτι και για την τιμή της θεωρίας. Μου είπαν ότι από, τον, από το Φεβρουάριο η θεώρηση θα κοστίζει 80 ευρώ. Εγώ νομίζω ότι στην πράξη αυτό δεν αποτελεί διευκόλυνση, το αντίθετο θα έλεγα. Είναι επιβάρυνση και ε, προσπάθεια να δυσκολευτεί η χορήγηση τέτοιων θεωρήσεων. Οπότε ίσως θα έπρεπε και η εκτολιστική εξουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επανεξετάσει το θέμα αυτό. Μήπως θα έπρεπε να γίνουν κάποιες εξαιρέσεις, σε πάση περιπτώσει, για αυτού του είδους ε, της ε, Νομίζω ότι δεν είναι κατάλληλο το επίπεδο των 80 ευρώ. Ευχαριστώ. Άλλοι ομιλητές. Έχουμε εκπρόσωπο της ε, Κομισιόν ή της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης μαζί μας. Όχι, ε. ε συνήθως έρχονται, γι' αυτό ρωτάω. Μήπως είναι εδώ και φοβούνται να πάρουν το λόγο. Παρακαλώ, παρουσιαστείτε. Έχουμε ερωτήσεις να σας, απευθύνουμε, να σας απευθύνουμε. 60, 80 ευρώ, ποιος είναι υπεύθυνο. Μπορείτε να απαντήσετε εσείς γι' αυτό. okay. Αν δεν θέλει ή δεν μπορεί η Κομισιόν, ο Πέτρας έχει το λόγο. Ε. Ναι, δεν έχουμε από ό,τι φαίνεται, Επιτροπή και Συμβούλιο, Πρόεδρε αλλά μιας και μιλάμε για διευκόλυνση θεωρήσεων και όχι απελευθέρωση, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και για το πρώτο βήμα τουλάχιστον, και για τις δύο πλευρές, φαίνεται να είναι αρκετά όσα έχουν γίνει και η τιμή που έχει συμφωνηθεί από τους Λευκορώσους είναι 3,5-35 ευρώ όταν αρχίσει να ισχύει η συμφωνία. Είναι σημαντική μείωση. Ακόμη και 35 ευρώ βέβαια είναι ένα σημαντικό ποσό για τους Λευκορώσους όπου ο μέσος μισθός δεν ξεπερνά τα 300 ευρώ. 35 ευρώ λοιπόν για όσους λάβουν θεώρηση βάσει των κανονισμών που θα εγκρίνουμε προσεχώς και θα έχουν δικαίωμα παραμονής στις χώρες που έχουν εφαρμόσει τη συμφωνία για 90 συνεχόμενες ημέρες σε ένα συνολικό διάστημα 180 ημερών. Τόσο μπορούν να μείνουν στην ευρωπαϊκή πλευρά. Και επίσης, Πρόεδρε, να αναφερθεί ότι η συμφωνία αυτή δεν θα ισχύσει στο βασίλειο της Δανίας, στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Με αυτές τις εξαιρέσεις πιστεύω μπορούμε να εγκρίνουμε τις συμφωνίες και η τελευταία μου παρατήρηση γιατί πήραν πέντε χρόνια διαπραγματεύσει με τη Λευκορωσία, αυτή την πλευρά να τη θέσουμε και στις δύο πλευρές, ιδίω στην ομάδα του Μίνσκ. που προσπάθησαν να διαπραγματευτούν κάποιε διατάξει που δεν ήταν ε, αποδεκτέ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουμε πιο δημοκρατική προσέγγιση. Ευχαριστώ, Πέτρα. Μόλι έμαθα ότι η κυρία από την ΕΕΔ μπορεί να θέλει να λάβει το λόγο. Πείτε μα το όνομά σα. Το όνομά μου είναι Ρόγκουλε, είμαι θυματάρχης για, το θέμα της Λευκο... για τα θέματα της Λευκορωσίας στην ΕΕ και να πω απλώς ότι λάβαμε ακριβώ το ίδιο αίτημα από τις λευκορωσικές αρχές, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να δούμε τη δυνατότητα να παγώσουν τα τέλη για τη θεώρηση στα 60 ευρώ. Αύριο ξέρουμε ότι στο Συμβούλιο θα υπάρξει ομάδα εργασία για τις θεωρήσεις στο Συμβούλιο και μετά από τη συνάντησή τους θα ξέρουμε ίσως περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό. Πάντως, Προς το παρόν η συμφωνία αξιοποιεί όλες τι δυνατότητε που αφήνει η συμφωνία και ο κώδικας για τι θεωρήσεις τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, άλλα σχόλια. Ωραία. Χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι τον Φεβρουάριο. Στις 3 Μαρτίου η ψηφοφορία στην Επιτροπή και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια αναμένεται να επιβεβαιωθεί. Όπως είχα ανακοινώσει, δεν έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Βαλμέιντα. Άλλη φορά θα γίνει αυτό. Οπότε πάμε στη συνάντηση των συντονιστών. Παρακαλώ, μόνον όσοι έχουν δικαίωμα να παραμείνουν στην αίθουσα να παραμείνουν